Ε, είναι μια δραστηριότητα που πρέπει να σταματήσει διότι έχουμε ήδη πολύ αρσενικό. Έχω τελειώσει με την έκθεσή μου, ελπίζω να μην ξεπέρασα το χρόνο. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο και θα ήθελα να ζητήσω να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά αναμένοντας ε, ε, την λήψη αποτελεσματικών μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης. Ευχαριστώ. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο το μέρος και θα έπρεπε να μείνει τόσο καθαρό όσο και όμορφο είναι τώρα. Για το καλό όλων μας. Ωραία. Με ενημέρωσαν ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει φτάσει ακόμα. Οπότε δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως να ακούσουμε τους ευρωβουλευτές στο μεταξύ, να δούμε τι έχουν να πούνε. Αλλά βέβαια, αν δεν μπορεί να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μήπως να περάσουμε στην επόμενη. Μπορείτε, αγαπητέ κύριε, να περιμένετε λίγα λεπτά, ώστε να εξετάσουμε πρώτα την επόμενη αναφορά και μετά να επανέλθουμε στη δικιά σας. Μόλις έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Ωραία. Καλώς. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η αναφορά που έχει να κάνει με την γεωργία και την, βιο... την βιολογική γεωργία. Για τις μειώσεις των ενισχύσεων στην βιολογική γεωργία. Είναι εδώ οι αναφέροντες. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε. Καλησπέρα. Είμαι ο Αντρέ Γαρθία. Γεωργός στην βιολογική γεωργία και εκπρόσωπος της Unión de Uniones από την Καστίγια Λαμάντσα, μια οργάνωση των αγροτών. Συμμετέχω και στην οικολογική πλατφόρμα της Καστίγια Λαμάντσα και σας ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε για το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας έχει να κάνει με την αλλαγή στις διατάξεις όσον αφορά τις ενισχύσεις μέσω προγράμματος υπέρ της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Και αυτό δύο χρόνια τώρα. Παρόλο που έχουν υπογράψει τη σύμβαση για ενίσχυση πέντε χρόνια, υπό τον όρο θα συνεχίσουν βέβαια τις βιολογικές τους δραστηριότητε. Η διάταξη αυτή όμως ίσχυσε αναδρομικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι άλλαξε η κατάσταση στα μέσα του δρόμου. Και από πού που είχαμε 7% ενίσχυση, για 3.900 και αγρότες. Στις 5 Ιουλίου του 2014 η κυβέρνηση της Καθήγια Μάνσα έστειλε στην Επιτροπή το πρόγραμμα M11, Βιολογική Γεωργία, με ενισχύσεις που θα έδινε παρόμοιες με αυτές των προηγούμενων ετών. Στις 13 Νοεμβρίου του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε τις δικές της παρατηρήσεις. Καμία όμως δεν αφορούσε τις ενισχύσεις στις 27 Μαρτίου του 2015 η Περιφερειακή Κυβέρνηση δημοσίευσε τον νόμο βάσει του οποίου ορίζονται οι βάσεις για τις επιδοτήσει στη βιολογική γεωργία. Και εκεί αναφέρονται τα ποσά ενισχύσεων που υπήρχαν στο πρόγραμμα το οποίο είχε σταλεί στην Επιτροπή το 2014, χωρίς παρατηρήσεις. Καλή την πίστη λοιπόν και βάσει της ε, εμπιστοσύνη που είχαμε στην νομοθεσία του Μαρτίου 2015 και στο σχετικό πρόγραμμα ζήτησαν ενισχύσεις οι αγρότες για βιολογική γεωργία για πέντε χρόνια. Όμως η νομοθεσία λέει ότι δεν μπορεί να αλλάξει η βοήθεια αν δεν υπάρξει η έγκριση του προγράμματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είχε ελεύθερο το, το δρόμο η κυβέρνηση να αλλάξει τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις όπως θέλει, όσο θέλει, χωρίς να σεβαστεί την ε, σταθερότητα δικαίου, τη βεβαιότητα δικαίου. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2015 στάλει το πρόγραμμα στην Επιτροπή με τις διορθώσεις και φάνηκε ότι υπήρχε διόρθωση στις ενισχύσεις. 9 Οκτωβρίου του 2015 στάλει το πρόγραμμα προς έγκριση. Η περιφερειακή κυβέρνηση εγκρίνει τις διορθώσεις προκειμένου να αλλάξουν εντελώς οι ποσότητες των ενισχύσεων στη βιολογική γεωργία και μειώθηκαν μέχρι και 67% χωρίς καμία παρατήρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήταν ε, ε, στην αρχή έτσι όπως είχαν πάει στην Κομισιόν χωρίς καμία παρατήρηση. Και τώρα άλλαξαν. Οπότε εμεί δεν καταλαβαίνουμε γιατί η περιφερειακή κυβέρνηση άλλαξε το ποσότητε των ενισχύσεων, ενώ είχε ήδη συγκαλέσει την έναρξη του προγράμματος για τον Ιούλιο του 2014 ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει αναδρομικά την αλλαγή ενός προγράμματος που πλήττει την νομική βεβαιότητα. Ποιος τελικά προστατεύει τα συμφέροντα των Γιώργων. Στη συνέχεια, το Μάρτιο του 2016, η Περιφερειακή Κυβέρνηση δημοσίευσε τον νόμο τροποποιώντας αυτόν το 2015 για να μειώσει τις ενισχύσεις παρόλο που πριν από ένα χρόνο είχαν πέσει υπογραφές για την επόμενη πενταετία. Η Περιφερειακή Κυβέρνηση λοιπόν της Καστίγια Λαμάντσα αλλάζει αυθαίρετα τις ενισχύσεις όσο περνάει ο καιρός χωρίς καμία εξήγηση. Οπότε δεν υπάρχει πια καλή την πίστη. Η περιφερειακή κυβέρνηση υποφελήθηκε από την αλλαγή αυτή ώστε να δώσει 400 εκατομμύρια σε δασικές ε, περιοχές μέση της δημόσιας επιχείρησης Αθεκάν. Και έγινε μια νέα συμφωνία για τα δάση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως πρέπει να ελέγξει ότι δεν υπάρχει απάτη. Δεν έκανε όμως τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ε, τηρούνται τα του κανονισμού 303 του 13, το άρθρο 6 που αναφέρεται στη νομική βεβαιότητα για παράδειγμα, το άρθρο 8 που αναφέρεται στις περιβαλλοντικές συνέπειες, το 26 που μιλά για διαφάνεια στη διαδικασία, ενώ εδώ πέρα μας κρύψανε πληροφορίες. Το 29, βάσει το οποίο η Επιτροπή αξιολογεί το πρόγραμμα, βάζει παρατηρήσεις που θα έπρεπε να διορθώσει η Καστίγελα Μάντσα. Όμως έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή του προγράμματος του 2014, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε καμία απολύτως παρατήρηση όσον αφορά τα ποσά των ενισχύσεων, ούτε ζήτησε αναθεώρηση οποιαδήποτε αλλαγή. Άρθρο 30 που επιτρέπει την τροποποίηση μόνο εφόσον έχει εγκριθεί το πρόγραμμα και όχι πριν. Επίση, δεν τηρήθηκαν τα του κανονισμού του 2005 του 2013, το άρθρο 5 που μιλάει για καταστροφή του περιβάλλοντος και το άρθρο 11 που εφαρμόζεται μόνο εφόσον έχει εγκριθεί το πρόγραμμα και όχι πριν. Ενώ αυτά που έγιναν δεν δικαιολογούνται βάσει του άρθρου 11. Τέλος. Πιστεύουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών θα ανοίξει έρευνα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει, να δει γιατί επιτράπει μια αλλαγή σε πρόγραμμα και δέχτηκε τέτοια συμπεριφορά από τις αρμόδιες αρχές Κάτι το οποίο βέβαια θέτει σε κίνδυνο τη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας στην Καστίγια Ντελαμάτσα και ε, επιφέρει και κινδύνους όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Και με αυτό περνάμε στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν, τον κύριο Βόκιας και τον κύριο Έμπερχερτς. Μπορείτε να απαντήσετε και οι δύο όπως θέλετε. Μπορείτε να μοιράσετε το χρόνο σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε επανειλημμένως ε, με τον αναφέροντα. Έχουμε λάβει και μία ε, καταγγελία που έχει ταξινομηθεί και έχει λάβει ήδη απάντηση ο αναφέρον. Τώρα για το θέμα, η περιφέρεια της Καστίγια Λαμάντσα έχει δημοσιεύσει ήδη το μέτρο της βιολογικής ε, γεωργίας, ε, υπάρχει τέτοιο δικαίωμα, αλλά δικαίως ε, έθεσαν μια επιφύλαξη, λέγοντας ότι η δημοσίευση αυτή γίνεται υπό προϋπόθεση έγκρισης του προγράμματος. Η Επιτροπή μέχρι εκεί δεν συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση είναι κάτι το οποίο γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας, με ευθύνη της περιφέρειας. Η Επιτροπή λαμβάνει το πρόγραμμα και αφού λάβαμε το πρόγραμμα, το λάβαμε με τα ποσά ε, ε, στήριξης που θεωρεί μειωμένα ο καταγγέλων. Δηλαδή, ό,τι έχει γίνει μέχρι την υποβολή του προγράμματο είναι εσωτερικό θέμα τη περιφέρεια. Η Κομισιόν δεν συμμετείχε στη συζήτηση αυτή. Εμείς λάβαμε λοιπόν το πρόγραμμα με τα ποσά τα οποία ο καταγγέλων θεωρεί ε, μειωμένα. Το αίτημα λοιπόν του καταγγέλλοντος ε, γιατί η Κομισιόν ε, δεν αντέδρασε σε αυτή την αλλαγή δεν υπήρχε λόγος, δεν μπορούσαμε. Έγιναν συζητήσεις κατά τη διαπραγματεύση του προγράμματος, έγιναν άτυπες διαπραγματεύσεις αλλά το τελικό πρόγραμμα περνάει πρώτα απ' όλα από μια εσωτερική συζήτηση στην περιφέρεια. Και η περιφέρεια βάσει τη δική τη στρατηγική, των δικών τη πολιτικών ζητημάτων, αποφασίζει ένα σύνολο μέτρων και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει μέσω ενό συνόλου μέτρων και αφού κάνει τη συζήτηση με όλου του ενδιαφέρουμενου τομεί, ε, συμφωνώντα και τα ποσά κατά μέτρο, καθώς και τα ποσά για την βιολογική ε, ε, γεωργία. Μας κοινοποιεί όλα αυτά και αφού γίνει αυτή η κοινοποίηση ε, της οριστικής, του οριστικού προγράμματος, τότε μιλάμε για το τρέχον ποσό. Δεν μιλάμε για μείωση της ενίσχυσης. Μιλάμε για το τρέχον ποσό, οπότε για την Κομισιόν δεν υπήρξε μείωση. Όλα έγιναν κανονικότατα και νομιμότατα. Ήθελα να σας δώσω και κάποια στοιχεία. Η Καστία Λαμάντσα, όταν υπέβαλε το πρόγραμμά της, παρουσίασε έναν προϋπολογισμό του οποίου το 14% ε, ήταν αφαιρωμένο στην ε, βιολογική ε, καλλιέργεια, βιολογική γεωργία, ενώ ο ευρωπαϊκός μας είναι 16%. Και όχι μόνο αυτό, η τελευταία τροποποίηση, δεδομένης μεγάλης ζήτησης που υπάρχει, με αυτό το μειωμένο ποσοστό που ε, αναφέρει ο καταγγέλων ε, υπήρξε ευρεία ε, εκτέλεση του προγράμματος από τις καλύτερες που είχαμε ποτέ στην Καστία Λαμάντσα, στην Ισπανία και πιθανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 28% του προπολογισμού αναλώθηκε ήδη πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι η διαχειριστική αρχή αύξησε και άλλο τον προπολογισμό και αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει το 15% του συνόλου του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης ποσοστό δηλαδή που έχει δεσμευτεί για την βιολογική καλλιέργεια, για τη βιολογική γεωργία, για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ζήτησης. Με ένα ποσό το οποίο καταγγέλλον λέει ότι είναι μειωμένο, έχουμε αύξηση της, ε, της ζήτησης ε, για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Αύξηση της ζήτησης συμμετοχή στο πρόγραμμα, Και τέλος θέλω να πω ότι για μας την Κομισιόν οποιαδήποτε αίτηση αύξησης ενός κονδυλίου ε, για ένα πρόγραμμα ε, μιας γραμμής δράσης σημαίνει ότι πρέπει να τα πάρουμε από κάπου αλλού. Ε, και υπάρχει μια ισορροπία την οποία πρέπει να τηρούμε ανα πάσα στιγμή και αιτιολογημένα μάλιστα. Έχουμε και άλλες αιτήσει. Έχουμε τους νέους γεωργούς που ζητούν αύξηση, τη δασοκομεία, κάτι πολύ επίκαιρο, υπάρχει αύξηση της ζήτησης σε πολλούς τομείς. Πρέπει λοιπόν η περιφέρεια ε, και η Κομισιόν να μπορέσουν να αιτιολογούν κάθε αλλαγή στον προπολογισμό. Και μόνο όταν υπάρχει πρόβλημα, για παράδειγμα, αν βλέπαμε ότι η ζήτηση των, για την, των γεωργών για τη βιολογική γεωργία μειώνεται, εκεί θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε το κατά πόσο τα ποσά είναι ε, κατάλληλα δεσμευμένα. Αλλά εδώ δεν είμαστε σε αυτή την περίπτωση. Ευχαριστώ. Ε, εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα ο λόγος στους συναδέλφους. Η κυρία Βαλίνα. Ευχαριστώ, Σεσίλια. Από την περιοχή αυτή, αλλά και αλλού στην Ήπεθρο, πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να υπάρχει στήριξη από τη δημοσιοδίκηση για αυτό το είδος παραγωγής, τη βιολογική που καταλαβαίνετε ότι έχει δυσκολίες, άρα χρειάζεται κάποια εγγύηση και για τις τιμές αλλά και για τα έσοδα των μικρών αυτών εκμεταλλεύσεων που αφιερώνονται στην βιώσιμη γεωργία. Σύμφωνα με τα όσα εγκρίναμε μάλιστα από ό,τι ήταν στην προηγούμενη Ολομέλεια για τις πατάλεις, τα τρόφιμα που πετάμε. Ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε μια δύναμη κατάσταση εξαιτίας των ε, πολιτικών των χωρών μελών και πολλές φορές και εξαιτίας και της αδιαφορίας των κυβερνούντων να προστατεύσουν τους μικρούς παραγωγούς και μερικές φορές ε, είναι τα θύματα ε, εμπορικών συμφωνιών τεράστιων που κάνουμε σε διεθνές επίπεδο. Η ιδεολογική γεωργία πάντως είναι ακριβώς αυτό το οποίο μπορεί να μας προστατεύσει στο μέλλον, το βιολογικό και προστατεύει και το περιβάλλον από την κλιματική αλλαγή. Άρα συνάδει με τόσα συμφωνήθηκαν στο COP21. Θα έπρεπε λοιπόν να στείλουμε μια επιστολή στις αρχές της ε, Καστίγια Λαμάντσα να μας εξηγήσει περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι κάτι το οποίο πλήττει πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δικιά της την πλευρά θα έπρεπε να μας εξηγήσει κατά πόσο η νέα και η νέα γεωργική πολιτική θεωρείται ότι δίνει περισσότερα χρήματα στις μονάδες εκείνες οι οποίες ε, κάνουν βιολογική καλλιέργεια. Θα ήταν ενδιαφέρον να το ξέρουμε αυτό. Ευχαριστούμε ε, ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους αναφέροντες που ήρθαν. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ξεκαθαρή απάντησή της. Πρώτον, πιστεύω ότι η αναφορά δεν έχει θέση εδώ, δεν είναι σωστή, δεν είναι κατάλληλη. Γιατί, γιατί έρχεται, προέρχεται μάλλον από μια εσωτερική συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή θέλει να καταστήσει ευρωπαϊκό ένα ζήτημα το οποίο είναι εσωτερικό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εμπλακεί σε αυτή την εσωτερική συζήτηση και είναι και άδικη γιατί ε, λένε ότι ζημιώνεται η οικολογική βοήθεια τη στιγμή που παίρνει το τριπλό κατά μέσο όρο περιοχή αυτή από την Ευρώπη για τέτοιες δραστηριότητες. Και έπειτα υπάρχει και θέμα διαδικασίας. Πολύ καλά τα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της. Ισχυρίζονται οι αναφέροντες ότι μειώθηκαν οι ενισχύσεις βάσει ενός ε, διατάγματος σε δύο μήνες διαφορά από κατεκλογές τοπικές, λέγοντας ότι υπήρξε μείωση σε σχέση με το τελικό πρόγραμμα. Αυτό όμως που δεν υπολόγισαν είναι ότι το διάταγμα αυτό στο οποίο αναφέρονται προηγείται της έγκρισης του προγράμματος περιφερειακής ανάπτυξης. Μα οι ενισχύσεις αυτές δεν δίνονται, δεν αποφασίζονται αν δεν έχει εγκριθεί προηγουμένως ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό έγινε έξι μήνες μετά το διάταγμα του 2015. Και γνώρισαν ότι ανέφερε το διάταγμα αυτό την ρήτρα που έλεγε ότι τα μέτρα, τα προγράμματα, οι ενισχύσεις που καθαρίζονται δεν μπορούν να ε, προχωρήσουν αν δεν έχει εγκρίνει στο μεταξύ το πρόγραμμα η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι γίνεται μετά? Πρώτον, δεν υπάρχει εγκεκριμένο πρόγραμμα επίσημο, άρα δεν ε, υπάρχει κανένα δικαίωμα σε ενισχύσεις. Το δεύτερο είναι ότι το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης εγκρίνεται 6-7 μήνες μετά από το καθορισμό των πρώτων ενισχύσεων και φαίνεται ότι με τα εκτάρια τα οποία δικαιούνται ενισχύσεις λείπουν 160 εκατομμύρια. Οπότε τι κάνει η νέα περιφερειακή δίκηση, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων 40-50 εκατομμύρια ευρώ νομίζω προκειμένου να μπορέσουν ε, να δοθούν ενισχύσεις όλα τα εκτάρια που τη δικαιούνται, μειώνοντας τις ενισχύσεις ανεκτάριο εκτάριο, για να επωφεληθούν περισσότεροι. Οπότε καταλήγουμε να έχουμε το τριπλό σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη σε ενισχύσεις. Έπειτα πρόκειται για μια αυτόνομη περιφέρεια η οποία πάρα πολύ γρήγορα προχωράει στη χρηματοδότηση και βοηθάει και περισσότερους αγρότες που ζητούν αυτήν την ε, οικολογική ενίσχυση. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα υπαίθρου περιλαμβάνει και άλλα μέτρα εξυγχρονισμού ε, προς νέους γεωργούς, γεωργοί κτλ. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε εδώ με μια καταγγελία η οποία είναι καθαρά περιφερειακού χαρακτήρα και δεν ζημιώνει καθόλου κανέναν γιατί δεν είχε ακόμα εγκριθεί το πρόγραμμα αυτό περιφερειακής ανάπτυξης. Και θα τελειώσω λέγοντας ότι εδώ δεν συζητούμε το πόσο σημαντική είναι η οικολογία ή όχι, εννοείται όλοι συμφωνούμε ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό ότι όλες οι αρχές ευρωπαϊκές, περιφερειακές, τοπικές κτλ. πρέπει να την υποστηρίξουν. Εδώ πέρα μιλάμε για το αν υπήρξε ζημία από ένα περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο δεν είχε εγκριθεί εκ των προτέρων. Και αν τηρούνται οι κοινοτικέ διατάξεις ή όχι. Πέρα λοιπόν από την εσωτερική συζήτηση που γίνεται σε κάθε αυτόνομη περιφέρεια, δεν μπορούμε να πούμε ότι παραβιάζεται οποιαδήποτε ευρωπαϊκή διάταξη. Συνεπώ, εκ μέρου των σοσιαλιστών ζητώ να κλείσει η αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. το λόγο. Ε, Συμφωνώ με αυτά που είπε η Βελίνα από την Ισκέρδα τη συναδερφό μου, και στηρίζω και τους αναφέροντες. Κοιτάξτε, από τότε που βρίσκομαι εγώ εδώ σε αυτή την επιτροπή, τρία χρόνια αντιπρόεδρος, 80% των αναφορών έχει σαν αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι δεν είναι αρμόδια. Εμείς όμως οι ευρωβουλευτές τα ψάχνουμε, όπως για τα μωρά που έχουν απαχθεί, όπως για το ατύχημα στο μετρό της Βαλένθια και ένα σωρό άλλα περιβαλλοντικά και άλλα θέματα. Συνεπώς δεν είναι επιχείρημα σοβαρό αυτό. Εντάξει, είπε τη θέση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά εμείς έχουμε τη δικιά μας άποψη που μερικές φορές δεν ταυτίζεται με αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι εννοώ. Είναι αλήθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η κοινοτική πληροφορία είναι το πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό σκέλος και λειτουργούν βάσει της κοινοποίηση του προγράμματος αυτού που αναφέρει κάποια νούμερα, ποσά και τελείωσε. Ναι, αλλά οι κοινοί θνητοί που ζουν από τη Γεωργία στην Καστίγια Λαμάντσα πριν από την έγκριση του προγράμματος αυτού είχαν ένα διάταγμα που αναφερόταν σε κάποιες ενισχύσεις, βασίστηκαν σε αυτές. Και όταν ξαφνικά μειώνονται κατά μέχρι και 67% αυτές οι ενισχύσεις, καταλαβαίνετε πόσο πολύ ζημιώνονται οι αγρότες γιατί έχουν κάνει επενδύσεις. Και ξαφνικά τους λέμε 67% λιγότερο. Επίσης το αναδρομικό, θα το λέω για σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εσείς εντάξει κινήστε από τη στιγμή που έχετε το πρόγραμμα. Εντάξει, στο μεταξύ έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε ότι αυτό φταίει το ότι άλλαξε η κυβέρνηση, στο ότι άλλαξαν ε, και τα μέτρα. Ναι, αλλά δεν φταίει ο αγρότης που άλλαξε η κυβέρνηση. Το ότι αναδρομικά άρχισε να ισχύει ο νόμος, αυτό είναι το περίπλοκο στην υπόθεση. Και το θέμα της διαφάνειας, στο οποίο αναφέρθηκαν οι αναφέροντες, εννοείται δεν έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει να κάνει με τη συζήτηση στο περιφερειακό επίπεδο. Αλλά αυτούς τους πλήττει τελικά. Σίγουρα το στίχημα υπέρ της βιολογικής γεωργίας πρέπει να είναι μόνιμο και η Καστίγια Λαμάντσα αποτελεί παράδειγμα. Και γι' αυτό ίσως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από την περιφερειακή κυβέρνηση περισσότερες πληροφορίες. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μας βάζει σε σκέψεις. Οπότε θα μπορούσαμε να στείλουμε μία επιστολή που να ζητάει από την περιφερειακή κυβέρνηση εντάξει όχι να θεσμευτεί σε τίποτα, αλλά να βάλει αυτό το θέμα σαν προτεραιότητα. Γιατί Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε εμείς εδώ και είναι και ρόλος μας να πιέζουμε ώστε να μπαίνει σαν προτεραιότητα αυτό το ζήτημα, μια που η Καστίγια Λαμάντσα είναι πρωτοπόρο στο θέμα της βιολογικής γεωργίας. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε στη θέση της κυβέρνησης, αλλά μη τι άλλο να στείλουμε αυτή την επιστολή στην Καστίγια Λαμάντσα για να δούμε πώς θα μπορούσαν να εξετάσουν αυτό το ζήτημα κάπως αλλιώς. Και σίγουρα να κάτσουμε να σκεφτούμε για την κοινή γεωργική πολιτική, η οικολογική γεωργία, πώς ε, αναβαθμίζεται στην ε, καινούργια κοινή γεωργική πολιτική, αναβαθμίζεται ή όχι. Ευχαριστούμε κύριο Στέρη Ευχαριστώ Συμφωνώ με τις δύο προλαλήσεις σας. Και ειλικρινά με εκπλήσει αυτό που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί εγώ δεν ήξερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άκουγα, ή την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ισπανίας. Με εξέπληξε. Εγώ νομίζω ότι άλλο ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλο η Περιφερειακή Κυβέρνηση. Το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμετέχει δεν μπορεί να οδηγήσει στο να λέει πως ε, ό,τι έγινε είναι νόμιμο. Το ότι δεν συμμετείχε είναι ένα πράγμα. Το αν είναι νόμιμο ή δεν είναι, είναι παράτυπο αυτό το οποίο έγινε στην Ισπανία, αυτό είναι άλλο. Και τελικά παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ενέκρινε την δημοσιονομική ισορροπία της περιφέρειας. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να στηρίξει δημοσιονομικές προτεραιότητες. Θα μπορούσε. Δεν το έκανε όμω, την ισορροπία στήριξε. Γι' αυτό λέω ότι με ξέπλυσαν αυτά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ λοιπόν με τις συναδέρφους για τις αλλαγές στα ποσά. Οι αλλαγές βλέπετε στα ποσά και κυρίως στους κανόνες του παιχνιδιού οδηγούν σε νομική αβεβαιότητα. Και οι Ρωμαίοι έλεγαν πάντοτε ένας νόμος δεν μπορεί να ισχύει αναδρομικά. Έτσι. Συνεπώς, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που δύσκολα ε, μπορούν ε, να συγκεραστούν θα έλεγαν μη τι άλλο να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και η περιφερειακή κυβέρνηση μη τι άλλο να μας εξηγήσει κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι αρκετά ξεκάθαρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώνω το κατάλογο ομιλητών που είχα για αυτή την αναφορά, οπότε θα δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Καρθία Βακουέρο. Δύο λεπτά παρακαλώ ή ένας από τους δύο ή μοιραστείτε το. Ευχαριστώ. Η Καστίγια Λαμάντσα το 15% βάζει στην βιολογική γεωργία, είπατε. Και για το κλίμα. Μα το κλίμα είναι εξαιρετικό και μπορούμε να έχουμε εντελώ 100% βιολογική γεωργία. Οπότε όλος ο προβολισμό θα μπορούσε να πάει στην βιολογική γεωργία. Ο συνάδελφος. Εγώ θα προσπαθήσω να απαντήσω πρώτα απ' όλα στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και λυπάμαι για αυτά που λες. 25 Ιουλίου του 2014 εστάλει το πρόγραμμα της περιφέρειας σε εσά με τα ποσά που αναφέρονται από την αρχή, δηλαδή από τον Ιούλιο του 2014 τα ποσά ήταν γνωστά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Οικολογική Γεωργία. 13 ε, Νοεμβρίου του 2014 στείλετε κάποιες παρατηρήσεις στην περιφέρεια και δεν λέγατε τίποτα για τα ποσά αυτά. Τα γνωρίζατε όμως συνεπώς. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο τον Οκτώβριο του 2015 όταν σας ήρθε το τελικό πρόγραμμα που θα έπρεπε να είχε διορθώσεις, μπαίνει η μείωση αυτή του 67%. Από την άλλη, όσον αφορά το 15%, στην πραγματικότητα τα χρήματα που θα πηγαίνανε στην βιολογική γεωργία ήταν ένα 9% στο σχέδιο του 14 και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη και ο αριθμός των εκταρίων και όλα για να υπάρχει σύγκριση. Τα 400 εκατομμύρια που πήγαν στα δάση θα πηγαίνανε στη βιολογική γεωργία. Και λυπάμαι κύριε Κουτιέρη που δεν συμφωνείτε με τις ενισχύσεις που δεν είναι ίδιες με αυτές που έδινε πριν η κυβέρνησή σας. Αλλά το, η ρήτρα αυτή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για να τροποποιεί η εκάστοτε κυβέρνηση τον νόμο όπως το κατέβει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, τώρα εξαρτάται από μένα το πώς θα κλείσουμε εδώ. Ευχαριστώ και τους δυο σας που ήρθατε μέχρι εδώ. Αυτό πρέπει να κάνουμε, πιστεύω, είναι να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά και αυτό έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας της Επιτροπής μας. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, θα στείλουμε μια επιστολή στην περιφερειακή κυβέρνηση της Καστίγια Λαμάντσα όπου θα επισημαίνουμε ότι η αηφορία είναι κάτι που μας απασχολεί και ότι η αηφορία της βιολογικής ε, ε, γεωργίας ε, είναι κάτι που εξυπηρετεί και την αντοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την διατήρηση των πόρων που έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω λοιπόν ε, ότι και οι συνάδελφοι θα συμφωνούν μαζί μου ότι αυτό, αυτή είναι η σωστή οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ναι, συμφωνείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Ε, μιλήσατε για το τέλειο κλίμα για τη βιολογική γεωργία. Είναι πιστεύω τέλειο κλίμα και για ανθρώπου. Οπότε πηγαίνετε πίσω στην Ισπανία που είναι τόσο πιο, το, πολύ πιο όμορφη από τι Βρυξέλλε και τους καλύτερους μας χαιρετισμού στην Καστίγια Λαμάντσα. you very much. And now let's, let's... Ευχαριστούμε πολύ. Ας περάσουμε τώρα... You know that the commission... Ξέρετε, η Κομισιόν εξακολουθεί να μην είναι εδώ για να απαντήσει στον κύριο Μπρούνη. Έπρεπε να είναι εδώ πριν από πολύ πολύ ώρα, αλλά δεν εμφανίστηκαν. Οπότε εδώ βρίσκομαι σε δύσκολη θέση. Διότι πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα για αυτή την αναφορά. Έχουμε κανένα νέο. Ξέρουμε, έχουμε ακούσει κάτι την Κομισιόν, τους πήραμε τηλέφωνο. Κύριε Μπρούνι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Επειδή ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ε, εξακολουθεί να μην έχει έρθει, θα δώσουμε το λόγο σε αδέλφους ε, να παρέμβουν ε, για την υπόθεση αυτή της μόλυνσης της λίμνης, της Μπολσένα και μετά θα συνεχίσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να σας κρατήσουμε να περιμένετε για τόση ώρα. Νιώθω πραγματικά ντροπή εκ μέρους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργανών, όχι από την Επιτροπή μου. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος και φυσικά θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας, ε, αλλά η Επιτροπή παρέλειψε την υποχρέωσή της να είναι παρούσα εδώ. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά να καλέσω τους συναδέλφους να πάρουν το λόγο. Έχω ένα κατάλογο μιλητών, νομίζω. Όχι. Η κυρία Εύη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα και εγώ θεωρώ ντροπή να έχει έρθει ο αναφέρον ε, σε αυτή την Επιτροπή για να ακούσει μια απάντηση ε, για την αναφορά του και η Κομισιόν να μην είναι εδώ. Και εγώ ντρέπομαι πραγματικά. Δεν έχει συμβεί ποτέ νομίζω. Τρία χρόνια που είμαι εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή αυτή, ουδέποτε μου έχει τύχει κάτι τέτοιο. Η αναφορά αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική αφορά μια λίμνη, τη λίμνη Μπολσένα, που είναι κομμάτι του δικτύου Natura 2000, ε, ύψης της οικολογικής ε, σπουδαιότητας ε, λόγω της βιοποικιλότητάς της. Είναι μια ειδική ζώνη διατήρησης, ζώνη ειδικής προστασίας, οπότε εντάσσεται στην οδηγία για τα σηκωτόπους και στην οδηγία για τα πτενά. Είναι προστατευμένη περιοχή που θα έπρεπε να προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Λέω θα έπρεπε, διότι δυστυχώς όπως βλέπουμε σήμερα αυτή η λίμνη και τα νερά της ε, βρίσκονται σε μια κατάσταση ε, δεινή. Μας υπενθύμισε μάλιστα ο αναφέρον πως το 2013 ξεκίνησε μια διαδικασία έρευνας, ένα EU pilot ε, σε σχέση με την επεξεργασία των λιμάτων, των αποβλήτων και αναρωτιέμαι, και αυτό θα ρωτούσα και την Κομισιόν αν ήταν εδώ, Ποιε ε, ε, ενημερώσεις μπορούσε να μας κάνει σε σχέση με την πρόοδο αυτής της διαδικασία ε, έρευνα. διότι όπω φαίνεται μέχρι σήμερα οι τοπικές και εθνικέ αρχές δεν έχουν κάνει τίποτα ή μάλλον ελάχιστα. Τα μέτρα διατήρησης που έπρεπε να εφαρμοστούν μέχρι στιγμής αποτελούν, δεν αποτελούν πραγματικότητα και με την ενημερώση που ακούσαμε από τον κύριο Αναφερόντα με το διπλασιασμό των επιπέδων του φωσφόρου στα ύδατα εντός ενός έτους ε, καταλαβαίνουμε πόσο κακή είναι η κατάσταση των υδάτων και μας δείχνει τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά την προστασία των υδάτων ουσιαστικά ε, και πώς ε, έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα των υδάτων στα κράτη-μέλη ε, ενώ υποτίθεται ότι θα βελτιωνόταν τους λόγους τους υπενθύμισε ο αναφέρον είναι πολύ διάφοροι λόγοι, η εντατική γεωργία, ε, τα αστικά λύματα αλλά και πολλά άλλα. Ε, όπως το σχέδιο της γεωθερμικής εγκατάστασης ε, για την οποία υπάρχουν της γεωθερμικής μονάδας για την οποία υπάρχουν πολλές εμβολίες οπότε επαναλαμβάνω το αίτημα να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά το Ιταλικό κράτος και τα κράτη-μέλη, σε αυτή την περίπτωση το Ιταλικό κράτος, έχουν ε, παρουσιάσει τα δικά τους ε, σχέδια διαχείρισης των ε, υδάτων τους, οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως αυτή τη στιγμή δεν έχει μια εικόνα των υδάτων στα κράτη-μέλη και ειδικότερα στην Ιταλία. Πιστεύω λοιπόν ότι απέχουμε πολύ από το να λέμε ότι προστατεύουμε μια λίμνη που αποτελεί ε, κομμάτι του Natura 2000 ε, με ύψιστη οικολογική αξία και που θα έπρεπε να προστατεύεται. Ενώ δυστυχώς σήμερα, κατά την άποψή μου, οι εθνικές αρχές ε, δεν, κάνουν, δεν επιτελούν το καθήκον τους. Ευχαριστώ. Yeah. I find it scandalous. Εγώ το βρίσκω σκανδαλώδες το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν είναι εδώ. Πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Μια, μιας από τις σημαντικότερες οδηγίες μας είναι πραγματικά σημαντικό να τηρείται αυτή η νομοθεσία προκειμένου να διαφυλάσσεται και ο σεβασμό προ τα όργανα και προ την Κομισιόν. Γιατί αν η Κομισιόν δεν ανταποκρίνεται στι υποχρεώσει τη, τότε είναι πρόβλημα για όλου μα. Και δεν είναι μόνο η Ιταλία και οι αναφέροντε που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Όλοι μα το αντιμετωπίζουμε, διότι αντιμετωπίζουμε όλοι μα αυτό το. αυτού του είδου τα προβλήματα παντού. Ξέρετε, αντίστοιχα προβλήματα ε, έχουμε και στη Δανία και η κυβέρνηση της Δανίας επίσης αγνοεί και παραμελεί τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από την οδηγία για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. Αλλά δεν γίνεται να γίνεται μια τέτοια αναφορά, να υποβάλουμε ερωτήματα και στη συνέχεια να μην λαμβάνουμε απάντηση και να ελπίζουμε ότι ίσως κάποια στιγμή κάποιος μας απαντήσει για χρόνια. Άρα πρέπει να, ρωτήσουμε πολύ συγκεκριμένα την Κομισιόν, όχι μόνο το για ποιο λόγο δεν προσήλθαν σήμερα στη συνεδρίαση, αλλά τι σκοπεύουν να κάνουν προκειμένου να αποκατασταθεί και η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην ε, νομοθετική διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι, λέει η Πρόεδρος, το είπα και εγώ στην αρχή. Είναι πρωτοφανή αυτή η κατάσταση να μην ε, παρίσταται εδώ η Κομισιόν. Ε, προτού όμως ε, πούμε βαριά λόγια, ας αφήσουμε ένα μικρό ενδεχόμενο να έχει συμβεί κάτι σοβαρό. Διότι ε, στη δική μου θητεία τουλάχιστον είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί. Ας μην το, ξανααναλάβω, ε, ας μην το επαναλάβω λοιπόν. Θα ζητήσουμε εξηγήσεις από την Κομισιόν. Ενδεχομένως θα είναι πολύ δύσκολη η εξήγηση αυτή να δοθεί. Προφανώς άσχημα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά εγώ αναφερόμουν κυρίως στην, στην υπόθεση, στο περιεχόμενο της υπόθεσης που συζητούμε και εκεί δεν έχουν γίνει πολλά πράγματα. Αυτό είναι η, αλήθεια. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ. Εντάξει, λοιπόν, ε, ε, αναφέρθηκε ήδη ότι δεν είναι σωστό το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν βρίσκεται εδώ. Ε, θα ζητήσουμε εξηγήσει και γραπτές ή δυνατόν, προκειμένου να λάβουμε μια γρήγορη απάντηση από την Κομισιόν ε, διότι ε, εδώ φαίνεται ότι ε, υπάρχει μια καταγγελία ότι παραβιάζονται ευρωπαϊκές οδηγίες. Αν πράγματι είναι έτσι, τότε θα πρέπει η Κομισιόν να ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάση ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια συζήτηση, ένας διάλογος με το εκάστοτε κράτος μέλος. τα, έχουμε συζητήσει αυτά τα θέματα πολλές φορές. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι θα πρέπει να μείνει η αναφορά αυτή ανοιχτή και να λάβουμε το συντομότερο δυνατό της απαντήσεις της Κομισιόν. Φυσικά το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε ανοιχτή την, ε, την αναφορά. Το σημαντικότερο καθήκον μας βεβαίως είναι να συμβάλλουμε στην επίλυση του προβλήματος διότι είναι γεγονός ότι η ποιότητα του νερού ε, επιδεινώνεται, χειροτερεύει ε, διαρκώς, υπάρχει μια πτωτική, μια φθήνουσα πορεία γι' αυτό και ε, πρέπει σε κάθε περίπτωση ε, να το συζητήσουμε και με την Κομισιόν αυτό το θέμα. Εννοείται να αφήσουμε ανοιχτή την, ε, την αναφορά και εφόσον ε, λάβουμε την απάντηση της Κομισιόν να δούμε τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Ε, ευχαριστώ Πέτερ, ο κύριος Ταμπουράνο. Ναι, και εγώ συμφωνώ με όλες τις διαμαρτυρίες που ακούστηκαν για αυτό το να παράληψη. Ελπίζω να ελπίζω τέλος πάντων να είναι σοβαρός ο λόγος ε, ε, της απουσίας τους. Όσον αφορά τη λίμνη Μπολσένα, μέσα στα χρόνια η κατάσταση δεν ε, βελτιώθηκε, αντιθέτως επιδεινώθηκε. Εγώ θέλω να επισημάνω πόσο μεγάλο είναι ο κίνδυνο να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση αυτή. Εμεί έχουμε μια αρχή μα αρέσει πολύ, η αρχή τη ε, προφύλαξη. Ο Δόκτωρ Μπρούνι υπογράμμισε ήδη πόσο μεγάλο είναι ο κίνδυνο ε, επιδείνωσης της ποιότητας των υγρών εφόσον ε, οικοδομηθεί μια γεωθερμική μονάδα που παίρνει τα υγρά και τα ξαναρίχνει ε, δύο χιλιόμετρα μακριά στο κομμάτι το οποίο τροφοδοτεί τη λίμνη. Ε, μιλάμε για τεράστιες ποσότητες υγρών Και υπάρχουν μελέτες που επιβεβαιώνουν ότι δύο περιοχές ε, της ε, ε, λήψης των υδάτων και της απόθεσης των υδάτων επικοινωνούν, αλλά δεν υπάρχει επιστημονική άποψη ομόφωνη. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Εάν αυτές οι ζώνες δεν επικοινωνούν, οι μαλλιπικοινωνούν θα έχουμε τεράστιες επιπτώσεις για 25 χρόνια διότι αυτές οι... έχει δοθεί για 25 χρόνια. Μπορεί λοιπόν να δημιουργηθεί ε, πρόβλημα με τις γεωγραφικές ροές, ε, με ε, δηλητήρια από το αρσενικό, θα βρεθούμε ενώπιον μιας περιβαλλοντικής καταστροφής που γνωρίζουμε ήδη και Όλη η Ευρώπη, όλο ο κόσμος έχει ακούσει την καταστροφή του σεισμού της Αματρίτσε και εδώ έχουμε μια σεισμογενή περιοχή μεταξύ Ούμπρε και Λάτσιο. Αυτό λοιπόν μπορεί να οδηγήσει σε σεισμική δραστηριότητα τεχνητή που θα προσθεθεί στην φυσική και θεωρώ ότι οι κάτοικοι της κεντρικής Ιταλίας δεν χρειάζεται να εκτίθενται σε κινδύνους ε, τέτοιους ε, ανθρωπογενεί. Ζητώ λοιπόν η αναφορά να παραμείνει ανοιχτή ε, μέχρι να ολοκληρωθούν οι περαιτέρω έρευνες. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να κλείσουμε πιστεύω. Θα στείλουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις ε, που θέσατε στην Κομισιόν και θα τους ζητήσουμε γρήγορα, ε, θα, θα πω άμεσα μάλιστα, να μας στείλουν γραπτές απαντήσεις. Και τι απαντήσει αυτέ κύριε Μπρούνη θα σα τι στείλουμε το συντομότερο δυνατόν μόλι τι λάβουμε. Και φυσικά θα διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα ζητήσουμε από την Κομισιόν όπως επισήμανε ο Πετριγιάρ ε, ποια είναι η πρόθεσή τη. αν δεν έχει πρόθεση να ξεκινήσει η διαδικασία παραβάση για την υπόθεση αυτή διότι πρόκειται για μια πολύ ε, σοβαρή υπόθεση και σας διαβεβαιώ κύριε Μπρόνη εμείς το θέμα αυτό το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά στην Επιτροπή μας και θα θέλαμε να εκφράσουμε και το σεβασμό μας προς εσάς που χωρίς να είστε ένας άνθρωπος ε, υπερβολικά νέος ε, μπήκατε στον κόπο να έρθετε στις Βρυξέλλες ε, για να μας παρουσιάσετε όλη αυτή την, περι... την κατάσταση και την περιοχή με επιστημονική τεκμηρίωση που τεκμηριώνει ε, πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ λοιπόν σε εσά. Ε, εκτιμάμε ιδιαίτερα τι προσπάθειε που έχετε καταβάλει και τι συνεχεί προσπάθειε που καταβάλλετε ε, όσον αφορά τη Λίνδιν Μπολσένα. Ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε εδώ και σίγουρα θα δοθεί συνέχεια σε αυτό. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν. Και όπως ξέρετε, όπως έμαθα, ο κύριος αυτός είναι 90 ετών. Μιλάμε μερικές φορές για ανθρώπους που συνταξιοδοτούνται στα 65 και ο κύριος αυτός στα 90 το ασχολείται με ένα τόσο περίπλοκο ζήτημα. Ας τον χειροκροτήσουμε, πιστεύω, αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να επιστρέψετε καλά στο σπίτι σας. Ωραία. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο 8 αναφορά 0541 εξ ονόματος του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών για το πρόγραμμα βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Ο αναφέρον είναι ο κύριος Ευάγγελος Σιωμπανίδης. Είναι παρόν, είναι εδώ μαζί μας, ελπίζω. Σας χαιρετίζω θερμότατα. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Βρίσκομαι σήμερα στη δυσάρεστη θέση να καταθέτω κατά, στην Επιτροπή Αναφορών κατά της χώρας μου. Την παρούσα αναφορά που έχετε στα χέρια σας την καταθέσαμε πριν από δύο χρόνια και κάποιους μήνες αν θυμούμε καλώς. Μέχρι σήμερα που εξετάζεται η αναφορά η ελληνική κυβέρνηση ακόμα δεν έχει πληρώσει τους παραγωγούς. Τις τελευταίες μέρες ξεκίνησε να πληρώνει εκκρεμότητες του 2012. Το 2014 στους περι... σε όλους δεν έχει πληρωθεί. Σας έστειλε ο κύριος Αποστόλου, ο Υπουργός Γεωργίου της Ελλάδος, μια απάντηση που είπε ότι δεν πλήρωσε τους παραγωγούς διότι η χώρα μας είχε κάποιο πρόβλημα με τους βοσκοτόπους και ότι αν πλήρωνε θα έπρεπε να λάβουν μικρότερα ποσά από αυτά που τους αναλογούσαν. Από εκεί και πέρα, το ερώτημα είναι το εξή. Ο παραγωγός σε τι ευθύνεται πάνω σε αυτό. Ο παραγωγός, ο οποίος πληρώνει τους μελετητές, πληρώνει τους γεωπόνους, πληρώνει βιολογικές ζωοτροφές για να ταΐσει τα ζώα του και όλα αυτά τα χρόνια μένει απλήρωτος από το πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας. Όπως επίσης, δεν είπε ούτε λέξη, δικαιολογείται για τη μη πληρωμή τη βιολογική κτηνοτροφία με αυτά τα οποία λέει. Δεν μα είπε όμω, γιατί δεν πληρώνει και το πρόγραμμα τη βιολογική γεωργία. στην οποία δεν υπάρχει πρόβλημα βοσκοτόπων. Δυστυχώ, τα τελευταία χρόνια, από την εποχή που η Ελλάδα μπήκε στα μνημόνια και μετά, έχουμε να κάνουμε με μια απολωτρίωση όλων των αποθεματικών των ταμείων, μαζί με αυτά και τα χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία προορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για του παραγωγού, με αποτέλεσμα ε, βαθιά μέσα τους όλοι οι Έλληνες παραγωγοί πιστεύουν ότι τα χρήματα τα οποία παίρνει η ελληνική κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούνται προς άλλες ανάγκες της χώρας. Είτε για να πληρώσει μισθούς, είτε για να πληρώσει συντάξεις, είτε να πληρώσει ε, μνημονιακές δόσεις και όχι για να πάνε στους πραγματικούς δικαιούχους που όπως βλέπουμε με το πρόγραμμα των βιολογικών έχουν καθυστερήσει 3, 4 και 5 χρόνια να πληρωθούν. Θεωρούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και θα πρέπει να βρεθεί κάποιο τρόπο ώστε να συνετιστεί η ελληνική κυβέρνηση. Σα ευχαριστώ. Και εγώ σα ευχαριστώ και θα ανοίγω το ο λόγο για όλου του συναδέλφου. To... Ποιο θέλει. Α, ε, μάλλον όχι. Πρώτα θα στραφώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βέβαια, λέει η Πρόεδρο. Στην κυρία Νικόλ Σιλιανίδου, παρακαλώ. Αγαπητή Πρόεδρε, εστάλει στην Επιτροπή σας προς εξέταση αναφορά αυτή στα τέλη του 2015 και ο Γενικός Διευθυντής για την Γεωργία απάντησε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 29 Απριλίου του 2016. Όπως εξήγησε ήδη ο αναφέρον, πρόκειται για καθυστερήσεις σε πληρωμές για το ελληνικό πρόγραμμα 2007-2013. Όπω αναφέρεται στην απάντηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ενήμερη για τι καθυστερήσει στην καταβολή των πληρωμών για αιτήσει βάσει του προγράμματο βιολογικής κτηνοτροφίας στο πλαίσιο του ελληνικού προγράμματο αγροτική ανάπτυξη και αυτό έχει να κάνει με το σύστημα αναγνώριση αγροτεμαχίων και τη δυσκολία προσδιορισμού των επιλέξιμων για πληρωμή περιοχών. Οι ελληνικέ αρχέ λοιπόν δεν προέβησαν σε πληρωμέ για να αποφύγουν ε, σε περίπτωση ε, αχριωστήτως καταβληθέντων ποσών, να μην πρέπει δικαιούχοι να τα επιστρέψουν αυτά. Πρόκειται εδώ για το δεύτερο πυλώνα της γεωργικής ε, πολιτικής και ε, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδαν με σελικές αρχές ότι έχουν εξετάσει τις καθυστερημένες πληρωμές προς τους δικαιούχους. Τώρα έχουν πληρωθεί όλε οι υποχρεώσει. Οι ελληνικέ αρχέ είπαν ότι όλε οι πληρωμέ παραμένουν για το 2015 και 2016, όπω επίση και άλλε πληρωμέ που εκκρεμούν από προηγούμενα έτη, επειδή έγιναν προσφυγέ για παράδειγμα, τώρα προχωρούν και θα ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη του Ιουλίου του 2017. Τέλο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το νομικό πλαίσιο για το δεύτερο πυλώνα τη κοινή γεωργική πολιτική ε, ανάπτυξη της υπαίθρου δεν προβλέπει προθεσμίες πληρωμής σε αντίθεση με τους κανόνες που ισχύουν για τις άμεσες ενισχύσεις βάσει του πρώτου πυλώνα. Συνεπώς δεν υπάρχουν οικονομικές συνέπειες για τις χώρες μέλη εφόσον καταβάλουν καθυστερημένα ε, τα κονδύλια στους δικαιούχους. Για να ευθυγραμμιστεί η κατάσταση μεταξύ των δύο πυλώνων και να πληρώνονται έγκαιρα οι αγρότες, αυτή η ιδιαιτερότητα του δεύτερου πυλώνα θα τελειώσει το 2018 έτσι όπως προβλέπεται βάσει των ρυθμίσεων της κοινή γεωργικής πολιτικής που έχουν να κάνουν για την προγραμμική περίοδο 2014-2020. Για την επόμενη χρονιά, το 2018, οι πληρωμές στους δικαιούχους πρέπει να γίνουν από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31 Ιουνίου της επόμενης χρονιάς, όπως ισχύει για τον πρώτο πυλώνα. Η Επιτροπή δουλεύει πάνω σε πρόταση για τον εφαρμοστικό κανονισμό της Επιτροπής για υπολογισμούς πληρωμών σε δικαιούχους χωρών νομελών όταν πρόκειται για πληρωμές που καταβάλλονται μετά την προθεσμία. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι βάσει της κοινή ζωικής πολιτικής οι χώρες μέλη όταν αποζημιώνονται από δικαιούχους έτσι κι αλλιώς δεν τα παίρνουν πριν από τους ίδιους τους δικαιούχους. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος ευρωβουλευτής που θέλει το λόγο. Παρακαλώ, κυρία Κούνεβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, παρότι που δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με την αγροτική πολιτική γενικά και το προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων στο τομέα αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι όλη την Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τη βιολογική ανάπτυξη, τη βιολογική παραγωγή και πρέπει να έχουμε ένας προγραμματισμός συγκεκριμένο και η χρηματοδότηση η οποία τα λάβουν αυτοί οι άνθρωποι να είναι με ορισμό και να ελέγχεται από την Κομισιόν ή από την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης στο, Αγροτικής Ανάπτυξης. στο Ευρωκοινοβούλιο. Ε, όσο καταλαβαίνω, εδώ κάπου χάνεται κάποια χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσουμε έλεγχο. Και προτείνω να μην κλείσει η αναφορά, να την ελέγξουμε καλύτερα και αφού ξεκαταρίζουμε όλη η υπόθεση πώς έχει γίνει και έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση των ανθρώπων που παλεύουν με την βιολογική καλλιέργεια, τότε να την κλείσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πίτερ. Ευχαριστώ πολύ. Οι αναφέροντες εδώ παρουσίασαν ένα παράδειγμα για το πώς δεν πρέπει να ασκούμε πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχει ένας δεύτερος πυλώνας στη γεωργική πολιτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και σχετικά γενναιόδορη, γιατί αφήνει στα χέρια των χωρών μελών, στο δεύτερο πυλώνα, το τι θα κάνουν με αρκετά μεγάλο περιθώριο λιγμών. Αυτό όμως που συμβαίνει εδώ τώρα, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να υποσχόμαστε στους αγρότες ένα πρόγραμμα και μετά να μην τους πληρώνουμε. Πρέπει τα προγράμματα να προετοιμάζονται καλά, σωστά και να είναι έτοιμε και οι χώρε μέλη να πληρώνουν. Αλλιώ αυτό που κάνουμε είναι δυσφήμιση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε καθαρά. Δεν φταίμε εμεί Φταίει η χώρα μέλος. Ναι, αλλά από την άλλη κατάλαβα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να ρυθμιστεί το ζήτημα. Άρα δεν είναι δυνατόν να προσφέρονται προγράμματα στους αγρότες και μετά να μην πληρώνονται. Συνεπώς προτείνω να μείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή και επιπλέον να πάει στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Γίνεται τώρα τριμερής διάλογος για το όμνιμπους όπως γνωρίζουμε. Το πακέτο δηλαδή ελέγχου της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής προκειμένου να βελτιωθεί. Και το θέμα που συζητάμε εδώ έχει να κάνει με το Omnibus. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, άρα ας φροντίσουμε. Έτσι δεν είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά τουλάχιστον. Γιατί μας είπατε ότι μέχρι τον Ιούλιο του 2017 πρέπει να ολοκληρωθεί η ιστορία αυτή. Έτσι. Και μετά τι γίνεται. Διακόπτονται οι πληρωμές. Οι μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα πόσες είναι. Γνωρίζουμε το ποσό. Τέλος πάντων πρέπει να λυθεί αυτό. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί έτσι οι περιφέρειες και τα κράτη-μέλη δεν μπορεί να μην, να μην έχουν την ε, δυνατότητα να καταρτίζουν επιτυχημένα προγράμματα και χωρίς να καταβάλλονται τελικά τα, ποσά στους δικαιούχους. Το ερώτημα λοιπόν προς την Κομισιόν είναι ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Πόσες ε, πληρωμές δηλαδή εκκρεμούν ακόμη συνολικά. Ευχαριστούμε Πίτερ. Άλλος κανείς. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να απαντήσει τον Πίτερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκα στον Ιούλιο, γιατί αυτή είναι η πληροφορία που μας έδωσε η ελληνική κυβέρνηση στην απάντηση που έστειλε στην Επιτροπή Αναφορών στα τέλη Ιουνίου. Και αυτή είναι και η πληροφορία που έχουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ελληνικές αρχές δηλαδή λένε ότι θα ολοκληρώσουν τις παλιές πληρωμές που εκκρεμούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Και είπαν επίσης ποια είναι τα ποσά στην επιστολή των ελληνικών αρχών δηλαδή λέει ότι για τη βιολογική γεωργία ήταν περίπου 122 εκατομμύρια που μένουν να πληρωθούν και για την κτηνοτροφία 42,5 εκατομμύριο για τη βιολογική κτηνοτροφία. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστούμε. Καλώς. Ε, η πρόταση είναι η εξή βάση των παρεμβάσεων Θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή. Θα στείλουμε επιστολή στο Υπουργείο Γεωργίας εκφράζοντας την ανησυχία των ε, Ευρωβουλευτών βάσει των όσων μας παρουσίασαν οι αναφέροντες και όπως είπε ο Πίτερ. Θα παραπέμψουμε το θέμα και στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω πώς θέλετε να παρέμβετε πάλι οι αναφέροντες ή συμφωνείτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, είμαι ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη και ελπίζω ε, να βρεθεί κάποτε μια λύση σε αυτό το αιώνιο πρόβλημα που ταλανίζει τους Έλληνες παραγωγούς. Pues, eh, así es. Καλώς. Ωραία. Εφόσον συμφωνούμε, έτσι έχουν και τα πράγματα. Επιστρέφω την Προεδρία στην Πρόεδρό μας, η οποία επέστρεψε. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ ε, ε, που, που με βοηθήσατε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Χρειάστηκε να μείνω λίγο μόνη μου. Επόμενο θέμα. Με χαρά δίνω το λόγο στον ε, κύριο Ζόλταν Τόθ για να μας παρουσιάσει την αναφορά του. Είναι εδώ, είναι παρόν. Ελπίζω. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά bizottság elnökségét, a, a petíciós Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ την Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών και τους Ευρωβουλευτές μέλη της, αλλά και όλους τους παρόντες σήμερα εδώ. Θέλω να σας ενημερώσω σχετικά με, με ένα νέο στοιχείο. Γνωρίζετε βεβαίως την ε, ε, αναφορά μου, όπου σας ε, είχα περιγράψει και την τεχνολογία σχετικά με τις ρητίνες. Τι λοιπόν διαπιστώθηκε. Διαπιστώθηκε ότι ε, σε ορισμένα είδη μελιού που προέρχονται από την Ασία χρησιμοποιείται μία ε, μεθοδολογία, μια μεθοδολογια ρητινών μέσω της οποίας οποίας ε, φιλτράρονται ε, κατάλοιπα ε, φυτοκτόνων και αντιβιωτικών. Τέτοιου είδους προϊόντα λοιπόν έχουν εμφανιστεί και στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι προϊόντα τα οποία ε, καταστρέφουν μάλιστα και επιτίθενται ευθέω κατά των συμφερόντων ε, των Ευρωπαίων μελισσοκόμων και όχι μόνο αυτό, αλλά θέτουν αυτά τα προϊόντα και την, σε κίνδυνο την υγεία 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Ακριβώς διότι στα προϊόντα αυτά τα μελισσοκομικά παραμένουν κατά κατάλοιπα ε, φυτοκτόνων ε, και ε, αντιβιωτικών. Και μάλιστα δεν προστατεύεται κανείς με το να προμηθεύεται μέλι από δικό του μελισσοκόμο διότι ε, μιας και εφαρμόζεται αυτή η τεχνολογία ο κίνδυνος υπάρχει παντού και σε όλα τα προϊόντα. Πρόκειται στην ουσία για ε, δούριο ύπο. Ε, καθώς ε, ε, εμφανίζονται, διατίθεται στην αγορά προϊόντα τα οποία έχουν φίλτραριστεί με αυτή τη μεθοδολογία, με αυτή τη νέα τεχνική που χρησιμοποιείται στην Ασία και μάλιστα καθαρίζεται πλέον, φιλτράρεται με αυτήν την ε, μέθοδο και το κερί των μελισσών ε, μέσω μιας διαδικασία, μια διαδικασία μέσω της οποίας ε, μπορούν να μεταφερθούν τέτοιοι ρήποι και στο μέλι. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να ξαναπώ, να επαναλάβω ότι πρόκειται για έναν κίνδυνο για την δημόσια υγεία που αφορά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Στην πραγματικότητα έχουμε ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας δηλαδή και όχι μόνο στενά του κλάδου των μελισσοκόμων. Υποβάλαμε λοιπόν αυτήν την αναφορά για το μέλι, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι με αυτήν την ε, μεθοδολογία ε, ρητίνης παράγονται και μια σειρά από προϊόντα ζάχαρης. Ξέχασα δυστυχώς την, ε, τις διαφάνειες, την παρουσίαση που είχα ετοιμάσει. Παρ' αυτά, ε, αν πάτε στο Google και κάνετε μια αναζήτηση με τους όρους μέλη και ρητίνη, θα δείτε ότι είναι χιλιάδες τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε ε, έναν παραγωγό ο οποίος χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία ρητίνης ε, μέσω αυτής της εγκατάστασης που βλέπετε εδώ στη φωτογραφία. Και βλέπετε μάλιστα και τα διάφορα εργαλεία και τους διάφορους κάδους που χρησιμοποιούνται. Ως... Ε, ε, ε, επιστήμονα στον τομέα των τροφίμων πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να, χρησιμοποιηθούν, να χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους εργαλεία. Ακριβώς γιατί υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης και μάλιστα χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα κλειστό κύκλωμα τεχνολογίας. Ένας βιοαναλυτής λοιπόν ε, μπορεί να σας διαβεβαιώσει ότι ε, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί οι ορισμένες προϋποθέσεις να είναι ασφαλές αλλά κάθε ε, εργαζόμενος που ενδεχομένως δεν έχει τηρήσει τους κανόνες υγιεινής μπορεί να επιμολύνει μια τέτοια εγκατάσταση και στη συνέχεια να επηρεάσει αρνητικά το τελικό προϊόν. Δεν είναι δυνατόν να ε, αναμειγνύονται ε, ουσίες βενζολίου, στυρολίου ε, σε προϊόντα τα οποία ε, καταλήγουν στον Ευρωπαίο καταναλωτή ακριβώς γιατί είναι μεταλλαξιογόνα, καρκινογόνα πολλές φορές και γι' αυτό κύριοι Ευρωβουλευτές έχετε μια μοναδική ευκαιρία να δώσετε την δυνατότητα στους ε, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι βέβαιοι ότι ε, προστατεύεται η δημόσια υγεία και η προσωπική υγεία του καθενός. Γι' αυτό και το λόγο είναι απαραίτητο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται ε, σοβαρότατοι έλεγχοι ε, και να ελέγχονται όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα για στυρόλιο και βενζόλιο. Και, αυτό είναι και αυτή είναι και η ουσία του, της αναφοράς μας. Τέτοιοι έλεγχοι να γίνονται και στο μέλι και στο κερί. Επιδίωξή μου είναι λοιπόν, είναι σε κάθε έλεγχο να διερευνάτε και η παρουσία αυτών των καταλήπων. Ακόμα και στις δειγματοληπτικές έρευνες, στους δειγματοληπτικούς ελέγχους στα σούπερ μάρκετ. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Και αν, όπως είπα, ε, γκουγκλάρετε την ε, εταιρεία στην οποία αναφέρομαι και στην οποία ε, εντοπίστηκαν τα, προβλήματα είναι πραγματικά να σου σηκώνει τη τρίχα αυτά που διαβάζει κανείς εκεί στις ιστοσελίδες αυτές. Γιατί αν τα, αν τα τα στοιχεία αυτά θα δείτε ότι το μέλι αυτό ε, υπερθερμαίνεται και μάλιστα ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει και ένας κανονισμός του 2014 ο οποίος ορίζει ε, τα του μελιού ε, και με τροποποίηση αυτού του κανονισμού ε, θα μπορούσε να οριστεί ε, η υποχρέωση ελέγχου αυτών των μελισσοκομικών προϊόντων ώστε να εντοπίζονται συγκεκριμένα αυτά τα κατάλοιπα που σας ε, ανέφερα κατά την εισαγωγή αυτών των προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο για να μας διαφωτίσει. Παρακαλώ. Yes. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά να σας ε, δώσω την ε, οπτική γωνία της Επιτροπής. Η Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα για την ποιότητα του μελιού και έχει θεσπίσει νομοθεσία. Γι' αυτό ε, παίρνουμε λοιπόν πολύ σοβαρά αυτή την αναφορά, διότι όπως εξήγησε ο κύριος Τότ, η τεχνολογία αυτή όπως φαίνεται είναι δυνατή, οπότε παρακολουθούμε το ζήτημα είναι δυνατόν να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, ωστόσο, έχουμε ελάχιστα στοιχεία ότι πράγματι συμβαίνει αυτό. Έχουμε επικοινωνήσει και με την Ένωση Μελισσοκόμων ε, για να δούμε πώς μπορούσαμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες. Κάποιες πληροφορίες, κάποιες υποψίες ότι κάποια μέλια έχουν ε, πραγματι Προς το παρόν δεν έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίε. πληροφορίες. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν την πρωταρχική ευθύνη ε, για την επιβολή των κανόνων να το γνωρίζουν, τα ενημερώνουμε, αλλά πρέπει να γνωρίσουμε επίσης ότι οι τεχνικές ε, ανάλυσεις για τη διαπίστωση της παρουσίας της ρητίνης στο μέλι. Ε, δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολο να βρεθεί δηλαδή να εντοπιστεί αυτή η ρητίνη αυτού του είδους οπότε χρειαζόμαστε κάποια στοιχεία ε, για να ξέρουν και τα κράτη-μέλη που να ψάξουν. Τώρα, όσον αφορά το συγκεκριμένο υλικό το 859 που αναφέρθηκε στην αναφορά ως πιθανό ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτή την ε, δραστηριότητα δεν έχουμε ε, εγκρίνει φυσικά τη χρήση αυτή τη ουσία. έχει εγκριθεί να χρησιμοποιείται ως τροποποιητής ε, ε, για πλαστικά οπότε δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται αυτή η ρητίνη δεν ε, θα, ε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται με ασφαλή τρόπο αυτού του είδους ε, η ουσία. Και θα πρέπει να υπάρχει και νομοθεσία για τα κρατημέλη που να επιτρέπει στα κρατημέλη να δράσουν σε περίπτωση που εντοπίσουν αυτό το υλικό, αυτή την ουσία στο, στο μέλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τους συναδέλφους όπως εγώ που μερικές φορές βρισκόμαστε εμβρόντιτοι μπροστά στα όσα μαθαίνουμε διαβάζοντας αναφορές. Δεν είχα ιδέα ότι συνέβαιναν τέτοια πράγματα. Οπότε χάρη σε εσά πραγματικά μας διαφωτίσατε, μας μάθατε πολλά πράγματα. Τώρα ε, συνάδελφοι μπορείτε να έχετε τον λόγο πρώτο απ' όλο ο Πίτερ Γιάρ. Θα μπορούσε κανείς να πει σχεδόν ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σκάνδαλο που ε, εποάζεται αυτή την περίοδο. Λοιπόν, έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στην Επιτροπή Γεωργίας ε, το μέλι είναι δεδομένο για όλους μας ότι πρόκειται για ένα φυσικό προϊόν. Όποιος αγοράζει μέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι έχει αγοράσει ένα καθαρό, ένα φυσικό προϊόν. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο τη εμπιστοσύνη του καταναλωτή και ο καταναλωτή θεωρεί δεδομένο ότι αυτό το, το προϊόν που αγοράζει δεν έχει υποστεί επεξεργασία χημική. Ε, αν ε, αναφερόταν αυτό στη συσκευασία ότι πρόκειται για τεχνητό μέλι, τότε θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά σήμερα εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση κατά την οποία οι καταναλωτές θεωρούν δεδομένο ότι όταν αγοράζουν μέλι, αυτό το μέλι είναι φυσικό. Ε, τώρα υπάρχει κάποια διχογνωμία για το αν αυτό είναι βλαβερό ή όχι. Ε, η, όπως μας είπε η Κομισιόν ε, δεν επιτρέπεται αυτή η διαδικασία που μας περιγράφει εδώ ε, Δεν ξέρω. Από ό,τι ακούσαμε σήμερα εδώ, χρειάζεται να φωτιστεί το θέμα αυτό. Ε, διότι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα ακούσαμε σήμερα, ε, πρόκειται για σκάνδαλο. Ο καταναλωτής αγοράζει φυσικό μέλι και πρέπει να εξασφαλιστεί αυτή η εμπιστοσύνη ε, του καταναλωτή. Διότι ακριβώς ο καταναλωτή αγοράζει το προϊόν αυτό γιατί είναι φυσικό. Αλλιώ θα μπορούσε να φτιάχνει μέλι τεχνητά και μόνο στην κουζίνα του. Το αγοράζει όμως ακριβώς επειδή γνωρίζει ότι είναι φυσικό το προϊόν. Γι' αυτό και χρειάζεται να συνεχίσουμε την έρευνά μας στο θέμα αυτό, να το φωτίσουμε από όλε τι πλευρέ. Βλέπω, λέει η πρόεδρο, ότι γνέφεται καταφατικά. Νομίζω από την πλευρά μου ότι βέβαια θα σας δώσω το λόγο αν έχετε κάτι να προσθέσετε σε αυτά που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πίτερ Γιάρ. Οπότε καλύτερα πρώτα εσείς και μετά θα αποφασίσουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω ναι, να προσθέσω κάτι. Φυσικά θα περιοριστώ στα πέντε που έχω στη διάθεσή μου. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι στην Ευρώπη, εγώ ως αναφέρον για παράδειγμα, δεν είμαι υποχρεωμένος να ψάξω, να ερευνήσω και να έχω εγώ αποδείξεις που θα σας φέρω. Η ιδέα είναι να χτυπήσω το κουδούνι του συναγερμού, ώστε οι αρμόδιες αρχές, η αρχή των Ηνωμένων ας πούμε, κατάφερε να εντοπίσει αυτά τα στοιχεία μέσα σε προϊόντα. Τέτοια υπόλοιπα που έχουμε σε τρόφιμα εξαιτίας αυτής της τεχνολογίας ρητίνης. Και βρέθηκαν υπόλοιπα στυρολίου και βενζολίου. Συνεπώς, δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να φέρω αποδείξεις αλλά οι αρμόδιες αρχές να το ψάξουν και να βρούνε αν υπάρχουν τέτοια υπόλοιπα σε τιμές που δεν είναι επιτρεπτές. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι οι τιμές θα πρέπει να είναι μηδενικές, γιατί αυτές οι ουσίες είναι επικίνδυνες. Το στυρόλιο, ακόμα και στις πιο χαμηλές τιμές, προκαλεί εξέματα ή άλλους ερεθισμούς. Είναι γνωστό αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση βέβαια του καθενός μας διαφέρει. Αλλιώς εκτίθεται κάποιος ο οποίος δουλεύει μέσα σε ένα εργοστάσιο που επεξεργάζεται συμπολιμερές στη Ρόλιο και κάποιος άλλος που δεν δουλεύει εκεί φυσικά είναι εκτεθειμένος πολύ λιγότερο. Α, και κάτι ακόμα θέλω να ζητήσω στους ευρωβουλευτές να προτείνουν τροποποίηση του κανονισμού. Γιατί αυτό θα βοηθούσε πολύ τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι μία πρόταση λοιπόν για τροποποίηση του κανονισμού που θα μπορούσατε να υποβάλλετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι αναγκαίο κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και αν φαίνεται αστείο, ειλικρινά εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμμετάσχουμε σε ένα τέτοιο έργο μου, να εκπονήσουμε δηλαδή μια πρόταση τροποποίηση του κανονισμού. Ευχαριστώ, να σα βοηθήσουμε σε αυτή τη διατύπωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ ειλικρινά το βρίσκω φοβερό ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες η αρμόδια αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ενήμερη, έχει αναλάβει και δράση, ενώ η ΕΦΣΑ που είναι υπό τον έλεγχο της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν κάνει τίποτα, δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, ναι, κύριε Τσάκη, κόντευα να σας ξεχάσω γιατί αυτό το πράγμα πραγματικά με παθιάζει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να μείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, παρακαλώ, και να τη στείλουμε και στην Επιτροπή Γεωργίας. Να έχουμε και από αυτούς κάποια άποψη και μετά να αποφασίσουμε οριστικά. Πρόεδρος, δίκιο έχετε, σωστά. Ωραία προς ενημέρωσή μας λοιπόν. Θα στείλουμε την υπόθεση αυτή στην Επιτροπή Γεωργίας. Και στρέφουμε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν ακούμε συχνά ε, τόσο μεγάλες ανησυχίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από ό,τι κατάλαβα, ναι, εσείς θέλετε κάτι να κάνετε, γιατί ανησυχείτε κι εσείς και θα θέλετε να ερευνήσετε περισσότερο το τι συμβαίνει. Οπότε, σαφώς και θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά αυτή και περιμένουμε συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι σκοπεύει να κάνει. Για μένα θα πρέπει να αναλάβουμε δράση μαζί, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ωραία, παραμένει λοιπόν ανοιχτή αυτή η αναφορά και βασιζόμαστε στο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει συνέχεια και θα ενημερώσει και εμάς. Εντάξει. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε λοιπόν και που μας διαφωτίσατε για αυτό το θέμα. Εκ μέρους όλων μας, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που έχετε επενδύσει στην υπόθεση, που βρήκατε όλα αυτά τα στοιχεία. Σας ευχαριστούμε. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, Πρόκειται για την αναφορά 0978 σχετικά με την απαγόρευση των πλαστικών συσκευασιών για βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Η αναφέρουσα δεν είναι εδώ, αλλά έχει στείλει μια επιπλέον δήλωση και μας παρακολουθεί στο διαδίκτυο, γιατί αναμεταδίδεται η συζήτησή μας. Πρόκειται για την κυρία Βαντάστη, λοιπόν, αυτή είναι η αναφέρουσα. Θα κοιτάξουμε λοιπόν μαζί αυτή την υπόθεση. Πρώτα απ' όλα, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρακαλώ, η κυρία Λότς, να πάρει το λόγο και να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, αναφορά αυτή, που στην ουσία ζητεί την απαγόρευση των πλαστικών συσκευασιών στα τρόφιμα, και συγκεκριμένα στα φρούτα και στα λαχανικά και ακόμη πιο συγκεκριμένα από ό,τι καταλαβαίνω στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά. Εμείς ε, κάναμε τις παρατηρήσεις μας αναφερόμενοι αφενός στην ισχύουσα οδηγία για τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών που είναι και το σχετικό εργαλείο ε, που ε, διέπει την διάθεση συσκευασιών προϊόντων που διατίθεται στην αγορά και εκεί υπάρχει μια ιεράρχηση ε, των στόχων, που είναι πρώτον η πρόληψη των αποβλήτων, δεύτερη προτεραιότητα είναι η ανακύκλωση κτλ. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη μέσω αυτής της οδηγίας καλούνται να προλαμβάνουν τη δημιουργία αποβλήτων, την ανακύκλωση την, ε, των ε, αποβλήτων. Ε, από εκεί και πέρα όμως ορίζονται και το τι επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και τα πλαστικά επιτρέπονται. Υπάρχουν ορισμένες απαιτήσει βεβαίω που περιλαμβάνουν και τον όγκο και το βάρος του αποβλήτου που, θα πρέπει, που όπως λέει το, η οδηγία θα πρέπει να είναι το, κατά το δυνατόν ε, μικρά προκειμένου να μειώνεται, να μειώνεται ο συνολικός όγκος των αποβλήτων. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες βάσει των οποίων να μπορούν να απογορευτούν οι πλαστικές συσκευασίες για τα τρόφιμα και ιδίως πρέπει να παρατηρηθεί ότι η συσκευασία δεν μπορεί να θεωρείται ε, ξεχωριστά από το προϊόν που συσκευάζει. Ε, και εδώ υπάρχουν οι κανόνες που αφορούν και την υγιεινή των, ε, των, τροφίμων ε, και την, τα απόβλητα τροφίμων. Άρα δεν μπορούμε να πούμε γενικά ότι ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η πλαστική συσκευασία στα τρόφιμα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση αυτό όπου είναι απαραίτητο και αυτό είναι κάτι που οφείλουν να το αξιολογούν και να το εκτιμούν και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Υπάρχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και από το νάβου σχετικά με την προσυσκευασία, τα προσυσκευασμένα τρόφιμα και τα τρόφιμα που συσκευάζονται στο σημείο πώληση, Πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλές πτυχές, αλλά δεν μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ενωσιακό επίπεδο να υπάρξει ε, μια γενική απαγόρευση της, ε, των πλαστικών συσκευασιών. Υπάρχουν και κάποιες πρακτικές παρατηρήσεις που κάναμε. Αν δείτε, για παράδειγμα, στα, τα, τα αγκούρια που πολλούνται στα καταστήματα με αυτή την πλαστική μεμβράνη, εδώ είναι κάτι και αυτό μάθαμε και από τις επαφές μας με τον κλάδο ότι ε, η συσκευασία αυτή ε, είναι ε, κατάλληλη για το χειμώνα για παράδειγμα γιατί βοηθά να διατηρούνται αυτά τα προϊόντα δεν ισχύει όμως απαραίτητα το ίδιο και για το καλοκαίρι. Όπως και να έχει, ε, στο πακέτο για την κυκλική οικονομία προβλέπονται μια σειρά από μέτρα που το πακέτο που ε, ε, εγκρίθηκε από την Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2015 ενισχύσαμε και επαναπροσδιορίσαμε στόχους σχετικά με τις πλαστικές συσκευασίε που προφανώς έχουν κάποια αξία και κάποια σημασία και στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης και ε, παρουσιάσαμε και μια γενική στρατηγική, ε, μάλλον θα παρουσιάσουμε μάλλον μια γενική στρατηγική σχετικά με τα πλαστικά έως το τέλος του χρόνου. Και εκεί θα δούμε πιο συγκεκριμένα τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με την ε, τήρηση ε, συγκεκριμένων απαιτήσεων για, τα, για τις πλαστικές συσκευασίε των τροφίμων. Εκεί μπορούμε να εξειδικεύσουμε κιόλα τους κανόνες και να αυξήσουμε ή δυνατόν και τον, ε, τον, τον το, την ανακύκλωση ε, ή την επαναχρησιμοποίηση πλαστικών συσκευασιών. Αυτά από την δική μας πλευρά, έτσι γενικά, ε, σχετικά με την αναφορά αυτή και βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στους συναδέλφους, κύριε Χόκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή. Σας παρακολουθώ εδώ καιρό ε, έχουμε στοιχεία ότι βελτιώνονται τα προϊόντα. Μου έκανε έκπληξη που έμαθα ότι για τις μπανάνες, για παράδειγμα, που μου έκανε εντύπωση όταν το είδα, έχει βελτιωθεί η συσκευασία. Πρέπει να γνωρίζουμε όμως ε, τι υπάρχει μέσα σε αυτά τα πλαστικά. Και εκεί συνδέεται αυτό με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, γιατί και ε, εκεί μιλάμε για πλαστικά και η Κομισιόν ουσιαστικά έχει αποφύγει οποιαδήποτε σοβαρή αξιολόγηση των ενδοκρινικών διατρακτών όπως είδαμε πρόσφατα. Εκεί θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε λοιπόν τη δική μας έκκληση για πιο ασφαλή πλαστικά διασφαλίζοντας ότι όχι απλά θα μπορούν να επαναχρησιμοποιούνται και να ανακυκλώνται αλλά και ότι θα είναι καθαρότερα και δεν θα είναι αυτά που θα έπρεπε να είχαν αποκρευτεί εδώ και καιρό από την Κομισιόν. Η τα χημικά, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη αυστηρότητα και να δούμε πώς θα μπορέσουμε τι θα κάνουμε στο βαθμό που χρησιμοποιούνται τόσο πολλά πλαστικά σε επαφή με τα τρόφιμα. Αναφέρατε τα αγκούρια, αλλά ξέρετε μπορεί, να περάσουν οι ουσίες ε, μέσα στα ε, λαχανικά μέσα από το περιβλημά τους ε, ζητάμε πιο ασφαλή ε, συσκευασία αλλά εγώ θα έλεγα ότι η απαγόρευση των πλαστικών συσκευασιών δεν είναι η καλύτερη ιδέα για να αποφύγουμε τις πατάλη που επίσης είναι πολύ σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλους ομιλητές στον καταλογό μου. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά αφού έχουμε τη συναδελφό μας που είναι η πρώτη αγωνίστρια για τις ε, πλαστικές σακούλες το κρατάμε λοιπόν υπόψη μας αλλά δεν είναι ε, τώρα τέτοιες ε, εποχές που μπορεί να επιβάλλει γενική απαγορεύση των πλαστικών συσκευασιών η Κομισιόν δεν αποτελεί θέμα που εξετάζεται αυτή τη στιγμή ως ενδεχόμενο ε, αλλά για να κάνουμε ένα βήμα με αυτή την αναφορά. Ε, θα ευχαριστήσω την ε, αναφέρουσα που έθιξε το θέμα και μας οδήγησε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και η Κομισιόν φυσικά θα συνεχίσει να εξετάζει τα ζητήματα αυτά και προς το παρόν έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες που έχει η Επιτροπή αυτή και μπορούμε να κλείσουμε την αναφορά σήμερα. Ωραία λοιπόν. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάμε στην τελευταία αναφορά για σήμερα, την 0108 σχετικά με τη θέση ψηδική επισήμανση για κρέας που παράγεται με τη χρήση μεθόδων εκτροφή που σέβονται τα ζώα και το περιβάλλον. Ο αναφέρον ο Χένιν Κράουζε δεν κατάφερε να είναι μαζί μας εδώ σήμερα, αλλά μας ε, παρακολουθεί μέσω web streaming. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την αναφορά σας και για τη συζήτηση που ανοίγεται σήμερα. Οπότε δίνουμε το λόγο στον κύριο Γκούμπελ, τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, απατώντας ε, στην αναφορά, να υπενθυμίσουμε το γενικό πλαίσιο τις επιλογές ε, ε, ε, επισήμανσης τρόφιμα σε σχέση με τον τρόπο παραγωγής. Πέραν από την επισήμανση για την ανθρώπινη κατανάλωση, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιβάλλει καμία υποχρέωση εναρμονισμένα στους παραγωγούς αντιθέτως υπάρχει δυνατότητα βάσει των κανόνων ε, του κανονισμού 69 του 2011 οι εκτροφείς να αναφέρουν ε, τέτοιες πληροφορίες εθελοντικά. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια. Η Κομισιόν φυσικά συνεργάζεται με τις αρχές των κρατών μελών όσον αφορά την αναρμονισμένη εφαρμογή της νομοθεσίας στα κράτη-μέλη και φυσικά επειδή το αναφέρει ο αναφέρον το ζήτημα της μεγαλύτερης εμπιστοσύνης στα συστήματα που επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές ή που οργανώνονται από τις δημόσιες αρχές σε αντίθεση με τα συστήματα που έχουν αναπτύξει οικονομικοί φορείς ε, δίνει λοιπόν και, υπάρχει λοιπόν και δυνατότητα για τα κράτη-μέλη να εισαγούν τέτοια συστήματα επισήμασης σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει μια διαδικασία κοινοποίηση, ε, συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, πρέπει να αποδείξουν ε, ότι ο στόχος του μέτρου είναι επαρκής προστασία των καταναλωτή, ότι υπάρχει ενδιαφέρον των καταναλωτών και ότι έχει νόημα να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος ε, να εφαρμόσουμε κάποιο υποχρεωτικό σύστημα ε, αναφοράς πληροφοριών που να αφορούν την ευημερία των ζώων για την παραγωγή κρέατος. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας ε, είναι αρκετά πιστικά. Θεωρούμε λοιπόν βάσει πολλών μελετών και εκθέσεων που έχουν γίνει για συγκεκριμένους τύπους κρέατος Έχουμε λοιπόν αποδείξει ότι αυξάνεται το κόστος της παραγωγής, ε, οπότε κάποια στιγμή θα υπάρξει και αύξηση του στιγμής για τους καταναλωτές το να εφαρμόσουμε μια τέτοια, το να υποχρεώσουμε μια τέτοια κάτι τέτοιο στους παραγωγούς ε, Επίσης έχουμε αποδεικτικά στοιχεία ε, για το τι είναι σημαντικό για τους καταναλωτές ε, όταν κάνουν τις επιλογές τους. Όταν βλέπουμε πληροφορίες που σχετίζονται με την ευημερία των ζώων ή τη βιωσιμότητα γενικότερα, δεν είναι Εμείς παράγοντες αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι κάποιοι άλλοι είναι πιο σημαντική. Βέβαια εξαρτάται από τι ομάδε των καταναλωτών, άλλοι είναι πιο διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα ε, αν αυξηθεί η τιμή για τέτοιους λόγους. Ε, οπότε θεωρούμε ότι η σημερινή επιλογή που έχουμε της ε, θελοντικής επισήμανσης είναι ο καλύτερο τρόπο, όπου οι παραγωγοί μπορούν να κάνουν και να προβάλλουν τις προσπάθειε που κάνουν επιπλέον των άλλων των συστημάτων που χρησιμοποιούν και κάποιοι καταναλωτέ μπορεί να ενδιαφέρονται να πληρώσουν αυτό το παραπάνω ποσό ώστε το κρέα που αγοράζουν να παράγεται υπό συγκεκριμένε συνθήκε. Ο αναφέρον ε, λέει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία που λένε ότι το επιπλέον κόστο δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και αναφέρει φυσικά και την υπόθεση ε, του συστήματος ε, του πίνακα για το σύστημα αυτό ε, που αναφέρει την ε, παραγωγή του Tablex. εκεί ξέρετε η κατάσταση είναι πιο απλή χρησιμοποιεί τα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ε, με κάποιους αριθμούς που ας πούμε επισημαίνονται πάνω στα αυγά στον τομέα του κρέατος υπάρχει άλλη προσέγγιση τα ζώα και τη διάρκεια της ζωής τους μπορεί να έχουν υποστεί πολλές διαφορετικές ε, συνθήκες διαβίωσης ε, οπότε θα ήταν πολύ πιο πολύπλοκο το σύστημα που θα μπορεί να απεικονίζει ακριβώς ποιες συνθήκες σε ποιες συνθήκες έζησαν Καταλαβαίνουμε φυσικά την έκκληση αυτή για την επισήμανση του νουπού κρέατος, αλλά θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του κρέατος παράγεται στην Ευρώπη, πηγαίνει σε επεξεργασμένα τρόφιμα. Οπότε είναι ακόμα αμφισβητήσιμο κατά πώς θα πρέπει να επιβάλλουμε ένα τέτοιο Ακριβώ σύστημα για το κρέα που αντιστοιχεί μόνο σε ένα κομμάτι τη αγοράς. Οπότε προ το παρόν δεν προτιθέμεθα να κάνουμε οποιαδήποτε πρόταση νομοθετική για αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αγκάθα Κρίστη μου θυμίζει η κατάσταση στην αίθουσα. Ένα ένα φεύγουν από την αίθουσα οι διάφοροι ευρωβουλευτέ. Έχω όμω τον Πίτερ που είναι ακόμα παρόν εδώ και εσά. Ναι, ακριβώ. Τώρα θα έπρεπε να ψηφίσουμε για κάτι πολύ σημαντικό, ε, έτσι. Εμεί θα αποφασίσουμε αν ψηφίζαμε τώρα, εμείς για όλου. Τέλος πάντων, δεν έχει ζητήσει εδώ κανείς το λόγο, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι με εμπιστεύεστε για να συνοψίσω, ε, ή όχι. Παρακαλώ, Πίτερ. Ναι, θέλω να πω ότι συμφωνώ επί της ουσίας με τη γνώμη που εξέφρασε η Κομισιόν. Αν θέλετε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλλονται πολλές προσπάθειες, πολλές φορές και από τους ίδιους τους γεωργούς, ε, προκειμένου να ε, δημιουργηθούν ε, πιστοποιητικά ή σήματα ποιότητες. Είναι λίγο σαν το αυγό του Κολόμβου, διότι σε κάποια προϊόντα μάλιστα υπάρχουν υπερβολικά πολλά σήματα ε, και είναι δύσκολο κανείς να διακρίνει τι τελικά ε, διατίθεται και τι όχι. Αν καταφέρουμε σε ορισμένα χρόνια να ενιοποιήσουμε κάπως το σύστημα, ίσως τότε θα μπορούσε να, τα πράγματα να γίνουν πιο απλά. Αυτή τη στιγμή ε, είναι δεδομένο νομίζω και συμφωνούμε όλοι ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια φάση αναζήτησης. Προσπαθούμε λοιπόν να διερευνήσουμε ε, πώς θα μπορούσαν να ενυποηθούν αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα πράγματα. Ε, νομοθεσία συγκεκριμένη δεν χρειάζεται. Ελάχιστες απαιτήσει, ελάχιστα πρότυπα, ε, βεβαίως, γιατί όχι. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ με την άποψη ότι αυτή τη στιγμή δεν απαιτείται η θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, διότι το ζήτημα μπορεί πολύ καλά να ρυθμιστεί σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Συμφωνώ και εγώ, είναι προαιρετικό ε, τα κράτη-μέλη ε, να ε, θεσπίζουν απαιτήσει σε εθνικό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια γενική υποχρέωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπω μα είπε η Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε τον αναφέροντα για το γεγονός ότι έθεσε το ζήτημα αυτό. Σας ευχόμαστε να περάσετε καλά σήμερα το βράδυ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και ε, συνάδελφοι καλό βράδυ και σε εσά. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας.